Να περάσουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Κύριε Πιτέλα, ζητήσατε το λόγο για την ημερήσια διάταξη. Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για τη διαδικασία που αφορά την εκχώρηση οικονομίας ε, της αγοράς ε, στην ε, Κίνα ε, το Συμβούλιο των Υπουργών ε, Μπορείου στα τέλη του Μαΐου θα συνεδριάσουν και μετά θα πάνε στην Ιαπωνία και τον Ιούλιο θα δοθεί συγκεκριμένο σημαντικός προσανατολισμός. Εμείς οφείλουμε οπωσδήποτε να έχουμε ε, το δικό μας σχέδιο λέγοντας από πλευράς μας ότι θα πρέπει να αποφευθούν αποφάσεις που θα ζημιώσουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και γι' αυτό προτείνω να ασχοληθεί το Κοινοβούλιο σήμερα με την ένταξη στην ημερήσια διάταξη μια συζήτηση και ψηφίσματο για το Κίνα. Δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να σιωπήσει ενώπιον μια υπόθεση που κινδυνεύει να ζημιώσει χιλιάδε χιλιάδων επιχειρήσεων και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεων απασχόλησης. Ποιος θα ήθελε να υποστηρίξει το αίτημα αυτό του κυρίου Πιτέλα. κύριος Μπορέλη. Ναι, σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ γιατί υπογραμμίσατε αυτό το θέμα. Εμείς είμαστε υπέρ, γιατί μάλιστα έχουμε υποβάλει το ίδιο αίτημα, το γνωρίζετε καλά, για τους ίδιους λόγους που υπογράμμισε και ο κύριος Πιτέλα. Περιμένουμε και οι υπόλοιπε ομάδε να στηρίξουν αυτό μα το αίτημα. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς να εκφραστεί κατά αυτού του αιτήματο. Παρακαλώ. Ο κύριος Κασπάρη. Κύριε Πρόεδρε, στην Ευρώπη, σε αυτή τη συγκυρία, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα ανησυχούν για τη θέση εργασίας τους. Και έχει να κάνει με το εάν θα δοθεί καθεστώς οικονομία της αγοράς και τι δυνατότητες θα δημιουργήσει αυτό. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να είμαστε λαϊκιστές. Θέλουμε να ασχοληθούμε ακριβώ με το μέλλον αυτών των εργαζομένων. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον κατέληξε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή κάνει την μελέτη αντικτύπου και τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μα υποβάλει μια πρόταση σε αυτή τη βάση. Σε αυτή τη βάση λοιπόν οι συντονιστέ έχουν ένα χρονοδιάγραμμα για την περαιτέρω αντιμετώπιση του θέματο αυτού. Και επαναλαμβάνω, το θέμα δημιουργεί πολλά συναισθήματα αλλά είναι και πολύ σημαντικό. Άρα το θέμα δεν είναι να υπάρξει κάποιο πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα, αλλά το μέλλον των εργαζομένων. Δεν χρειαζόμαστε τίτλους, χρειαζόμαστε σωστές λύσεις. Όχι λοιπόν ακτιβισμό, αλλά σωστή στάση και αποφασιστική κατά των ε, Κινέζων εταίρων μας. Σας παρακαλώ να αποσύρετε λοιπόν αυτό το αίτημα, να επιτύχουμε καλή συνεργασία. Σκεφτείτε τους πολλούς εργαζόμενους και όχι διάφορες προπαγανδιστικές ενέργειες. Θα σας ήμουν ευγνώμων να αποσύρατε αυτό το αίτημα. Ο κύριος Λάμπερτς. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω μια συμβιβαστική λύση. Νομίζω πως αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι μόνο συναισθηματικό. Είναι ένα θέμα πολιτικό, βιομηχανικό, είναι οικονομική πολιτική. Και αν το Κοινοβούλιο θέλει να εισακουστεί, καλό θα είναι να εκφράσει την άποψή του πριν από την Κομισιόν και όχι μετά. Εγώ λοιπόν ε, συμφωνώ με τα επιχειρήματα των σοσιαλιστών και του Έρντεντα για να γίνει πριν η συζήτηση. Όμω τίποτα δεν μα εμποδίζει να το κάνουμε αυτό στην πρώτη σύνοδο του Μαΐου στο Στρασβούργο. Είναι ήδη εντό χρόνου. Προλαβαίνουμε να οργανώσουμε σωστά τη συζήτηση και όχι να τη βάλουμε τελευταία στιγμή στην ημερήσια διάταξη και να προετοιμάσουμε και να προβλέψουμε και ένα ψήφισμα στο τέλο τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Λάμπερτ. Νομίζω ότι το αίτημα του κυρίου Πιτέλα. Παρακαλώ κύριε Πιτέλα. Ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την πρόταση του συναδέλφου Λάμπερτς με την προϋπόθεση ότι όντως η συζήτηση και το ψήφισμα θα γίνουν πριν από την, από την Κομισιόν. Δηλαδή στο Στρασβούργο θα γίνει συζήτηση και ψήφισμα. Δεν ψάχνουμε να βρούμε πρωτοσέλιδα, ούτε να κάνουμε προπαγάνδα. Θέλουμε, θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα και τα προβλήματα λύνονται όταν το Κοινοβούλιο εκφράζεται, όχι όταν σωπαίνει και δεν ψηφίζει τίποτα. Κύριε Μπορέλη. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εμείς συμφωνούμε με την πρόταση των Πρασίνων για τους ίδιους λόγους που εξέφρασε και ο κύριος Πιτέλα. Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Βέμπερ, εφόσον υπάρχει αυτή η συμβαστική πρόταση, θα ήθελα να υποβάλω το εξής αίτημα. Δεν θα ήταν δυνατόν να προπαρασκευάσουμε το θέμα αυτό στην επόμενη διάσκεψη των Προέδρων. Υπάρχει πριν από την προηγούμενη Ολομέλεια συνεδρίαση τη Επιτροπή των Προέδρων να δούμε πώ ακριβώ θα το αντιμετωπίσουμε στην Ολομέλεια του Μαΐου. Θα πρότεινα να ε, αποστείλουμε το θέμα στη διάσκεψη των Προέδρων. Πρόεδρο, ωραία. Λοιπόν, κύριε Πιτέλα, ζητήσατε να γίνει συζήτηση σήμερα και το ψήφισμα στην πρώτη ολομέλεια του Μαΐου. Αυτή δεν ήταν η αρχική σας πρόταση. Όχι, μπορεί να γίνει και συζήτηση στο Στρασβούργο, όχι απαραίτητο σήμερα, με την προϋπόθεση ότι το ψήφισμα όμως θα γίνει στο Στρασβούργο. Δηλαδή τη συζήτηση μπορούμε να την κάνουμε σήμερα ή στο Στρασβούργο. Κύριε Πιτέλα, ενδιαφέρον. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Επαναλαμβάνω. Η συζήτηση τώρα και το ψήφισμα στην Ολομέλεια του Μαΐου στο Στρασβούργο. Αυτή ήταν η πρότασή σας. Παρακαλώ, παρακαλώ, ηρεμήστε. Μα αυτή είναι η πρόταση του συναδέλφου Πιτέλα. Λοιπόν, κύριε Λάμπερτς, εσείς προτείνατε εναλλακτικά και τα δύο, και η συζήτηση και το ψήφισμα να γίνουν στο Στρασβούργο. Ο κύριος Μπορέλη μόλις είπε, συμφωνώ με την πρόταση των σοσιαλιστών και των πρασίνων. Αλλά αυτό περιπλέκει τα πράγματα, γιατί είναι δύο διαφορετικές προτάσεις. Γι' αυτό πρέπει να επιχειρήσουμε να διευκρινίσουμε την κατάσταση. Κύριε Πιτέλα, κύριε Πιτέλα, Πιτέλα ακούστε με. Πείτε μας παρακαλώ τι ακριβώς ε, ε, θέλετε, για να δούμε τι θα ψηφίσουμε. Παρακαλώ κύριε Πιτέλα. Εγώ συμφωνώ να γίνει συζήτηση και ψήφισμα μαζί στο Στρασβούργο. Ωραία. Αλλά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα από αυτού, γιατί είναι θέμα της διάσκεψης του Προέδρων πλέον. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα για την ημερήσια διάταξη της ε, Ολομέλης του Στρασβούργου. Δεν μπορούμε. Οι προτάσει με βάση τον κανονισμό για την Ολομέλεια καθορίζονται στη διάσκεψη των Προέδρων. Μπορείτε να κάνετε μια δήλωση προθέσεων, τη λαμβάνω υπόψη, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε σήμερα. Ε, σκεφτείτε το. Πιτέλα, άμα είναι έτσι, Πρόεδρε, ξεκινήσουμε τουλάχιστον τη συζήτηση σήμερα και θα υποβάλουμε ψήφισμα για το Στρασβούργο. Okay. Ωραία, λέει ο πρόεδρο. Μα κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε, παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, ακούστε με, ακούστε με. Έχουμε έναν κανονισμό. Γιατί έχουμε κανονισμό. Γιατί είμαστε 750 και 8 πολιτικές ομάδες. Δεν είναι δυνατόν να εργαζόμαστε όπως να είναι. Γι' αυτό, επαναλαμβάνω, η ημερήσια διάταξη τη Ολομέλεια για το Στρασβούργο δεν μπορεί να αποφαστεί σήμερα. Δεν το προβλέπει ο κανονισμό. Και γι' αυτό το λόγο, εάν συμφωνείτε ότι θέλετε να συζητηθεί στο Στρασβούργο, τότε είναι μια σύσταση προ τη διάσκεψη των Προέδρων. Και εκεί θα ψηφιστεί. Σας προτείνω λοιπόν ότι το σώμα θα προτείνει στην επόμενη συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων την επόμενη εβδομάδα λοιπόν να συζητηθεί στην Ολομένα του Στρασβούργου το θέμα του, της Κίνας και να υπάρξει και ψήφισμα. Ποιοι συμφωνούν παρακαλώ. Κατά παρακαλώ. Αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Λοιπόν. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο αίτημα των σοσιαλιστών. Κύριε Πιτέλα, ζητήσατε να υπάρξει δήλωση τη Επιτροπή και του Συμβουλίου για τι πρόσφατε εξελίξει στην Πολωνία και τι επιπτώσει του στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ω δεύτερο σημείο για την ημέρηση διάταξη μετά την έκθεση Πυρίνσκι. Θέλετε αυτό να τεθεί στην ημέρηση διάταξη. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ποιο θέλει το λόγο. Ο κύριο Γκερέρο επ' αυτού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στην τελευταία Ολομέλεια εγκρίναμε με μεγάλη πλειοψηφία ένα ψήφισμα. Στο ψήφισμα αυτό εκφράσαμε την ανησυχία μας για την ε, παραλυσία του Πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου που έχει σαν αποτέλεσμα να διακινδυνεύει το κράτος δικαίου και δημοκρατία. Ζητούσαμε λοιπόν να τεθούν σε εφαρμογή οι συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και συγχρόνως ζητούσαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε διαρθρωτικό διάλογο με την πολωνική κυβέρνηση. Όμως επικεντρωνόμασταν στα συνταγματικά θέματα. Υπάρχουν και άλλα στην πολωνική πραγματικότητα που μας ανησυχούν. Για παράδειγμα, αυτά που έχουν να κάνουν με τα μέσα ενημέρωσης και πιο συγκεκριμένα η νέα ενδεχομένως ρύθμιση για την άμβλωση όσον αφορά τα δικαιώματα δηλαδή της γυναίκας και όλα όσα έχουν να κάνουν με την παραγωγική, αναπαραγωγική υγεία. Η ομάδα μου θα ήθελε το θέμα αυτό να συζητηθεί σήμερα με ψήφισμα, να προσθεθεί δηλαδή στην ημερήσια διάταξη μετά από την έκθεση Πυρίνσκι, ως δεύτερο θέμα στην ημερήσια διάταξη τη σημερινή. Ποιος θα ήθελε να υποστηρίξει αυτό το αίτημα. Η κυρία Μπιόρκ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίρνει σοβαρά τις αξίες της, ε, το σεβασμό για τη δημοκρατία και για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν τμήμα τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να καταστήσει σαφές ότι αυτά τα δικαιώματα τα υποστηρίζει και στην πράξη παντού. Τα δικαιώματα των γυναικών όμως ε, απειλούνται και περιορίζονται όλο και περισσότερο και είναι θεμελιώδη δικαιώματα τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, να μπορούν να αποφασίζουν για το σώμα τους. Το δικαίωμα να αποφασίζουν εάν θέλουν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί ή όχι. Γι' αυτό χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος θέλει να μιλήσει κατά. Ο κύριος Λιγκούτκο. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω ότι αυτού του είδους πρωτοβουλία εξαρτάται από τα προνόμια των χωρών μελών. Δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολωνική κυβέρνηση με κανένα τρόπο δεν θα αλλάξει την νομοθεσία για την άμβλωση. Αυτό είναι κάτι που έχουμε επαναλάβει ξανά και ξανά. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ορισμένοι δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό. Επειδή είναι αλήθεια ότι στην Πολωνία γίνεται συζήτηση επί του θέματος αυτού. Συζήτηση στην οποία συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών και το ψήφισμα θα ζητούσε από την κοινωνία των πολιτών δηλαδή να μην αναμειγνύεται σε αυτό το θέμα. Ε, είναι απαράδεκτο, είναι αλαζονικό Επιτρέπεται η συζήτηση από όσο ξέρω ακόμα, δεν απαγορεύεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορώ να επιτρέψω να γίνει συζήτηση για τα θέματα αυτά. Σήμερα είστε πολύ ζωηροί και αυτό είναι καλό. Αλλά ε, πρέπει να τηρήσω τον ε, κανονισμό. Μου είπατε ότι θέλετε να κάνετε μια συμβαστική πρόταση. Με ανησυχεί αυτό. <laughs> Γιατί μπορεί να μας προκαλέσει τις χέρες. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ιντφελτ και μετά στον κύριο Κονθάλεθ Πόνς, αλλά μετά πρέπει να ψηφίσουμε. Παρακαλώ, κυρία Ιντφελτ. Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Η ομάδα μου στηρίζει την αρχή συζήτησης, ψηφίσματος για θέματα που μας απασχολούν. Δεν βλέπουμε όμως για ποιο λόγο να γίνει αυτό τώρα, δεν είναι τόσο βιαστικό, οπότε προτείνουμε να γίνει το Μάιο, τον Ιούνιο, το αργότερο. Θα ήθελα όμως επίσης να πω στον συνάδελφο ότι βεβαίως και η κοινοβουλευτική και η κοινωνία των πολιτών της Πολωνίας πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριος Γκονζάλης Πόντς. Ευχαριστώ για την ε, Πολωνία. Έχουμε συζητήσει με την ίδια την Πρωθυπουργό και πριν από ένα μήνα εγκρίναμε ψήφισμα στο Στρασβούργο και στο ψήφισμα αυτό λέγαμε ότι άπαξ και υπάρχει κάτι καινούριο θα έρθει η Επιτροπή να μα το πει. Η Επιτροπή δεν ήρθε να μας πει τίποτα. Τον Ιούνιο θα συνεδριάσει η Επιτροπή της Βενετίας. Δεν έχει συνεδριάσει ακόμα, τη δώσουμε χρόνο. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα καινούριο στοιχείο που να μας επιτρέπει να συζητήσουμε. Μόνο η ενότητα του σώματος θα πληγεί από μια τέτοια συζήτηση. Σήμερα ακούσαμε ότι πρόκειται για νέα θέματα όχι για νομοθεσία, αλλά για προθέσεις ενδεχομένως για νέα νομοθεσία. Μα τα κοινοβούλια ποτέ δεν συζητάνε πάνω σε προθέσεις. Και δεύτερον, η πολιτική στην οποία ε, αναφέρθηκε η σοσιαλιστική ομάδα είναι πολωνικό ζήτημα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει ποτέ να μπαίνει μέσα σε αυτά και δεν πρέπει και να προκαταλαμβάνει την εθνική συζήτηση. Είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι το Πολωνικό Κοινοβούλιο. Λυπάμαι. Κύριε Γκερέρο. Ευχαριστώ. Θέλω να πω στον κύριο Κοζάλε Σποτς ότι όντω δεν είμαστε το Πολωνικό Κοινοβούλιο, είμαστε όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ακριβώς επειδή είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να συζητάμε για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν προτείνουμε να αντικαταστήσουμε την πολωνική κυβέρνηση. Αυτό που προτείνουμε είναι να συζητήσουμε για θέματα τα οποία απασχολούν κοινή γνώμη και πολιτική σκηνή μετά από αυτά που είπε η Σόφια Ντεβέλτ και η ομάδα Άλντε, εμείς θα θέλαμε να συζητηθεί τον Μάιο το ζήτημα αυτό, το πολύ τον Ιούνιο και όπως είπε και στο προηγούμενο θέμα ο Πρόεδρος, έτσι και εμείς τώρα θα προτείνουμε στη διάσκεψη των Προέδρων να συζητηθεί και αυτό το θέμα σε μία από τις δύο επόμενες ολομέλειές μας. Ωραία, άρα αποσύρετε το έτοιμά σας. Εντάξει, και θα δούμε τι έτοιμα θα υποβληθεί από την ομάδα σας στη διάσκεψη των Πρόεδρων. Οπότε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Οπότε, σύμφωνα... Μα γιατί φεύγετε, γιατί φεύγετε. Δεν τελείωσα. Καλά, εντάξει. Καλά. Λοιπόν, σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες προτείνω τις εξής αλλαγές στην ημέρη διάταξη για την Πέμπτη. Η ψηφοφορία θα συμπληρωθεί με δύο θέματα. Έκθεση Λεμπρετών για την άρση ασυλίας του κυρίου Πιέχα και ψηφοφορία για το αίτημα της Επιτροπής Απασχόλησης για, για διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Θέλει κανείς το λόγο επ' αυτόν? Ωραία. Καθορίζεται λοιπόν ε, το πρόγραμμα εργασιών μας με συμμετοχή ολίγων συναδέλφων. Για το διαδικαστικό έχει ζητήσει ο συνάδελφος Καστάλντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα διαδικαστικό θέμα. Θυμίζω τα άρθρα 22 και 141 ε, του κανονισμού μας και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας και των συναδέλφων στο καθήκον του Προέδρου να καθορίζει το ρόλο και τις εξουσίες του σώματός μας σε κάθε πτυχή της πολιτικής ζωής και ιδιαίτερα όσον αφορά τις διοργανικές σχέσεις. Αύριο θα ε, συζητήσουμε για νιωστή φορά, συνάδελφοι, δηλώσεις του περασμένου Μαρτίου ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το συζητήσουμε και τέρμα, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε, δεν, δεν είχαμε το δικαίωμα ούτε το καθήκον να εκφράσουμε τη δική μας βούληση και πολιτική ευθύνη. Αυτές ε, οι δηλώσεις λοιπόν είναι μόνο κατά ε, στο όνομα, στην ουσία πρόκειται για συγκεκριμένε ανελημμένες υποχρεώσει που, ευρωπαϊκές, οι οποίε ήδη έχουν δρομολογηθεί. Πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία και κανονικά θα έπρεπε να έχει υποβληθεί στη διαδικασία έγκριση, πρώην άρθρο 218 τη συνθήκη. Άρα λοιπόν η γνωμοδότησή μα επ' αυτού δεν είναι μόνο επιχρεωτική αλλά και δεσμευτική και γι' αυτό προτείνω σε όλου του συναδέλφους και ειδικά σε εσά, Πρόεδρε να ε, δεχτείτε το αίτημά μα για μια διαδικασία ακύρωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαστηρίου στο όνομα της Δημοκρατίας. Υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ε, Κύριε Καστάλτο, ευχαριστώ. Σημειώνοντας τα πρακτικά αυτά που είπατε, υποθέτω ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Διάξεσης των Προέδρων θα ασχοληθούν με το έτοιμά σας. Θέλει κανείς άλλο το λόγο για διαδικαστικό? Όχι. Ωραία. Τότε να περάσουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης, έκθεση του κυρίου Πυρίνσκι για την ετήσια έκθεση 2014 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Χαιρετίζω τον πρόεδρο της ε, Τράπεζας Επενδύσεων, Βέρναρ Χόια, και τους συνεργάτες του. Καλώς ήρθατε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να δώσω το λόγο στον εισηγητή, ο κύριος Πυρίνσκι. Παρακαλώ.